Uh, uh, Γεια σας συνάδελφοι και παρακαλώ καθίστε. Ξεκινάμε βεβαίως με μια ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Γκίφερ Χόφστατ, τον διαπραγματευτή μας για τον Brexit και τον κύριο Έλμαρ Μπρόκ. Και βεβαίως το θέμα είναι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Είχαμε εκφράσει το ενδιαφέρον μας ε, πολλές φορές ε, ήδη. Ε, προσφάτως είχαμε μία δημόσια κρόαση για τον αντίκτυπο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου σε ζητήματα δημόσιας υγείας και ασφάλειας τροφίμων και κατέστη σαφές κατά τη διάρκεια της ακρόασης πως η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα έχει σοβαρό αντίκτυπο σε θέματα αρμοδιότητός μας. Και βεβαίως ακούστηκαν και διάφορα πράγματα. Συμφωνήσαμε ότι αυτά θα τα λέγαμε στους διαπραγματευτές μας και στον κύριο Μπαρνιέ και γι' αυτό ακριβώς ε, καλέσαμε τους κυρίους Μπροκ, Γκουαλτιέρη να έρθουν σήμερα στην συνάντησή μας. Γι' αυτό ζητήσαμε τον κύριο Φερχόφτατ να έρθει σήμερα να μας πει τι γίνεται στις διαπραγματεύσεις και ποια είναι τα επόμενα βήματα. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε και θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, για την πρόσκληση που απευθύνονται σε μένα και στον Έλμαρ και ευχαριστώ και την Πρόεδρο της Επιτροπής και την Επιτροπή ολόκληρη. για τα όσα μας είπατε για την ε, ομάδα η οποία ασχολείται με το Brexit. Πράγματα πάρα πολύ χρήσιμα όταν εγκρίναμε τα τρία ψηφίσματα, γιατί μέχρι στιγμής έχουμε τρία ψηφίσματα. Αν μου επιτρέπετε λοιπόν, θα ήθελα να κάνω την παρέμβασή μου σε δύο μέρη. Πρώτα, μια γενική προσέγγιση του τι κάνουμε και το τι προγραμματίζουμε για τους επόμενους μήνες και μετά, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να έρθω στα συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν ε, την Επιτροπή σας και να σας υποβάλω πέντε ερωτήσεις ε, κλειδιά στις οποίες πρέπει να απαντήσουμε κατά την άποψή μου στην επόμενη φάση των ε, διαπραγματεύσεων. Αυτό θα έλεγα εγώ. Πρώτα απ' όλα. Πρώτα απ' όλα ε, για τη γενική προσέγγιση, όπως ξέρετε εγκρίναμε ένα ψήφισμα στις 13 ε, Δεκεμβρίου. Το Συμβούλιο ενέκρινε την ε, κοινή έκθεση Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέγοντας ότι υπάρχει επαρκής πρόοδος στα τρία βασικά ζητήματα, τα ξέρετε, δικαιώματα των πολιτών, τα οικονομικά και το θέμα της Ιρλανδίας ε, και αυτό σημαίνει ότι μαζί Συμβούλιο και Κοινοβούλιο κατέληξαν ε, στο συμπέρασμα πως υπήρχε επαρκή πρόοδο, επαρκής ε, πρόοδος, επαρκή προ, Επαρκής πρόοδος δεν σημαίνει βεβαίως ότι επαρκή η πρόοδος, αλλά και βεβαίως ε, έχει σημειωθεί όπως είπα κάποια πρόοδος αλλά σαφώς ε, είναι μεγάλη ακόμα ενισχύα για τα δικαιώματα των πολιτών Έχουμε τις αρμόδιες επιτροπές, ΛΥΜΠΕ, Γιούρι και την Επιτροπή Απασχόλησης ε, που θα ασχοληθούν με την διαδικασία που θα ακολουθήσουν οι Βρετανικές Αρχές, διαδικασία η οποία θα τεθεί προς την προς ε, επικύρωση. Οπότε η διαδικασία πρέπει να είναι φιλική προς τους ε, πολίτες, γιατί ξέρετε, όταν οι αρχές λένε ότι μια διαδικασία θα είναι απλή, ε, δεν συμβαίνει αυτό κατά κανόνα. Κατά κανόνα σημαίνει το αντίθετο. Εμείς ως κοινοβούλιο είμαστε υπέρμαχοι των δικαιωμάτων των πολιτών και πρέπει εδώ πέρα να κάνουμε σωστή δουλειά. Λοιπόν, Αυτά έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Ε, τι γίνεται στο μέλλον. Υπάρχουν τρία πράγματα που πρέπει να γίνουν. Τρία θέματα που θα μας απασχολήσουν στο Κοινοβούλιο. Πρώτον, πρέπει να επισημοποιήσουμε την ε, έκθεση προόδου να την μεταφράσουμε σε ένα επίσημο κείμενο συμφωνίας. Δικαιώματα πολιτών, το οικονομικό και το Ιρλανδικό ζήτημα. Και βεβαίω υπάρχουν και άλλα ζητήματα πέρα από αυτά τα τρία. Το δεύτερο θα είναι η συμφωνία που θα πρέπει να επιτευχθεί πριν από τον Μάρτιο για την ε, μεταβατική περίοδο. Χρειάζεται μία μεταβατική περίοδος και βεβαίω ε, θα πρέπει να συμφωνήσουμε πριν από τον Μάρτιο το ποιο θα είναι το σύστημα και ποια θέση θα έχει το Συμβούλιο. Και το τρίτο στοιχείο μετά είναι μια συμφωνία, η αρχή των διαπραγματεύσεων από τον Μάρτιο, όχι από τώρα, τον Μάρτιο και μετά, για την μελλοντική σχέση που πρέπει να οδηγήσει σε μια πολιτική δήλωση, πολιτική δήλωση η οποία θα είναι ένα ξεχωριστό έγγραφο ή ένα παράρτημα, εμείς θεωρούμε ότι καλύτερο είναι ένα παράρτημα, που θα έχει την συμφωνία αποχώρησης. Ε, θα έχουμε λοιπόν δύο μέρη την ίδια την Συμφωνία Αποχώρησης με τα τρία βασικά ζητήματα, δικαιώματα πολιτών, Ιρλανδία και το οικονομικό, και μια συμφωνία για την μεταβατική περίοδο που θα αποτελέσει τμήμα της συμφωνίας. Και μετά θα υπάρχει ένα παράρτημα στην συμφωνία, πιθανότατα, που θα είναι μια πολιτική δήλωση για τις μελλοντικέ σχέσεις Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Όλα αυτά πρέπει να γίνουν μέχρι τον Μάρτιο. Δηλαδή αύριο ουσιαστικά πολιτικά μιλώντας. Αυτά πρέπει να γίνουν ε, και να ολοκληρωθούν σε εννέα μήνες. Εντάξει, εννέα μήνες γεννάς παιδί βέβαια, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι μας αρκεί εμάς. Πώς θα οργανωθούμε τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πρώτο κομμάτι για την συμφωνία αποχώρησης έχουμε την μετάφραση της έκθεσης προόδου σε μια συμφωνία αποχώρησης και εκεί ως Κοινοβούλιο θα δώσουμε ιδιαίτερο βάρος στην διαδικασία που θα ακολουθηθεί στα δικαιώματα των πολιτών, διαδικασία η οποία για εμάς είναι ένα στοιχείο κλειδί γιατί μπορούμε να εγγυηθούμε στους Ευρωπαίους στην Βρετανία και στους Βρετανούς ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα ίδια δικαιώματα μέχρι τώρα γιατί α, ε, βεβαίως το θέμα είναι το εάν θα έχουν ε, το καθεστώς αυτό είχαμε ένα κατοκεκριτημένο καθεστώς αλλά εάν είναι τόσο γραφειοκρατική η διαδικασία και είναι εφιάλτης να αποκτήσει κανείς αυτό το καθεστώς θα, δεν έχει και πολύ νόημα. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μια διαδικασία η οποία θα είναι αυτόματη, χωρίς ε, διοικητικό βάρος για τους πολίτες της Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα είναι το κλειδί. Το δεύτερο θα αφορά την μεταβατική περίοδο. Το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων στις 29 Ιανουαρίου θα εγκρίνει τις κατευθυντήρες γραμμές ε, της διαπραγμάτευσης για τη μεταβατική περίοδο. Εκεί πέρα η σχετική ομάδα του Κοινοβουλίου έχει γνωμοδοτήσει προς το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων για τις κατευθυντήριες γραμμές. Οι κατευθυντήριες γραμμές λένε κυρίως το εξής, ότι η μεταβατική περίοδος μπορεί να είναι μόνο η συνέχεια του κοινοτικού δικαίου, της τρέχουσας κατάστασης. Δεν θα διαλέγουμε τα όσα μας αρέσουν ε, και θα λέμε ναι μας αρέσει η Τελωνιακή Ένωση αλλά όχι η ενιαία αγορά ή από την ενιαία αγορά μας αρέσει η ελεύθερη διακίνηση αγαθών υπηρεσιών και κεφαλαίων αλλά όχι ανθρώπων. Πρόκειται για συνέχεια της ε, τωρινής κατάσταση τη Βρετανία με μία διαφορά. Δεν θα υπάρχει εκπροσώπηση του Ηνωμένου Βασιλείου στο Κοινοβούλιο, στην Κομισιόν, στο Δικαστήριο, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην Κομισιόν. Οπότε, ε, να πω δηλαδή ότι θα είναι μέλος χωρίς εκπροσώπηση. Αυτή θα είναι η μεταβατική περίοδος η νομοθεσία θα συνεχίσει να ισχύει, η πολιτική θα συνεχίσει να ισχύει, θα συνεχίσει να έχει τον τελικό λόγο το ΔΕΚ, αλλά δεν θα υπάρχει εκπροσώπηση του Ηνωμένου Βασιλείου ε, στα θεσμικά όργανα κατά την διάρκεια της μεταβατικής περίοδου. Και το δεύτερο σημαντικό θέμα είναι πως το νέο σύστημα για τους Βρετανούς πολίτες που ζουν στη Βρετανία θα ισχύσει μόνο μετά την αποχώρηση και μετά τη μεταβατική περίοδο, κάτι το οποίο είναι φυσικό άλλωστε. Θα ισχύσει η νέα διαδικασία μετά τη μεταβατική περίοδο. Κατά την διάρκεια της μεταβατικής περίοδου θα ισχύει το κοινοτικό κεκτημένο. Και αυτό είναι το τρίτο στοιχείο δηλαδή. Όταν θα τελειώσει η μεταβατική περίοδος, η πρόταση είναι να τελειώσει η μεταπατική περίοδος τον Δεκέμβριο του 2020. Το Κοινοβούλιο, όπως ξέρετε, ήταν κάπως πιο ανοιχτό ως προς αυτό και είχε πει πως θα μπορούσαμε να έχουμε τρία χρόνια ως περιθώριο. Λέμε λοιπόν στους διαπραγματευτές, ναι εντάξει να συμφωνήσουμε με το να τελειώσει η μεταβατική περίοδος τον Δεκέμβριο του 2020, αλλά μπορείτε να έχετε και κάποια ελαστικότητα όπως εμείς θεωρούμε ότι απαιτείται σε αυτές τις διαπραγματεύσεις και μετά. Το τρίτο θέμα που θα μας απασχολήσει θα είναι να διατυπώσουμε, σε, να διατυπώσουμε ένα νέο ψήφισμα που θα πάει στην Ολομέλεια του Μαρτίου. Ένα ψήφισμα λοιπόν το οποίο θα λέει το πώς βλέπουμε εμεί ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την σχέση μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχει τεράστια σημασία η Επιτροπή σας να μας ενημερώσει για τα πάντα, για οτιδήποτε αφορά την δημόσια υγεία, το περιβάλλον, την ασφάλεια των τροφίμων, οτιδήποτε αφορά είναι αρμοδιότητα της ΕΝΒΗ, γιατί θα είναι ένα αρκετά εκτεταμένο ψήφισμα. Έχει 16 παραγράφους. που θα δίνει μια γνωμοδότηση για τη μελλοντική σχέση. Έχουμε ήδη πει πως α, κατά την απόψή μας πρέπει να έχουμε μια συμφωνία σύνδεση σύμφωνα με το άρθρο 217. Αλλά θα έχουμε ένα κεφάλαιο που θα λέμε πώς βλέπουμε εμείς την εμπορική σχέση, την ε, θεματική συνεργασία. την συνεργασία σε ζητήματα εσωτερικής ασφάλειας ε, κτλ. Εξωτερική ασφαλείας ε, σε όλα αυτά. Στου τέσσερι πυλώνες που έχουμε. Για να το προετοιμάσω αυτό. Τι επόμενε ημέρε έχουμε κάποια σεμινάρια και κλεισμένων των θυρών με την Κομισιόν και κάτι παράλληλο κάνει το Συμβούλιο. Αυτό είναι το συνολικά το, το ζήτημα. Έχουμε τα 7 θέματα, συζητάμε την Κομισιόν και την ομάδα, την κατευθυντηρία του Brexit και έχουμε και τους πρόεδρους των Επιτροπών και τους συντονιστές των ομάδων που εκπροσωπούνται στην ε, ομάδα την κατευθυντήρια και έχουν εγκρίνει τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου. Ένα από τα 7 θέματα που συζητάμε και κλεισμένων των θυρών είναι πρώτον, κατόπιν που είναι πολύ σημαντικό για την ένβη, και θα προσκληθεί η ΕΝΒΗ αφορά το, τους ίσους όρους ανταγωνισμού, θέματα δηλαδή δημόσιας υγείας ε, και ασφαλείας ε, και θα ισχύσουν στο μέλλον. Θα λάβετε αυτή την πρόσκληση και με βάση αυτά τα σεμινάρια θα έχουμε ένα κείμενο που θα προετοιμάσει η ομάδα το οποίο θα στείλουμε σε εσά για να μπορέσετε να συζητήσετε το, το θέμα αυτό, τις δικές σας τις ε, επιθυμίες και το μελλοντικό ψήφισμα που θα εγκρίνουμε μέσα Μαρτίου. Και έρχομαι τώρα στο τελευταίο θέμα. Ποια είναι τα συγκεκριμένα ζητήματα εδώ. εντάξει, ε, κρούω ανοιχτέ θύρε. Δεν ξέρω αν το λέτε στα αγγλικά αυτό. Όσον αφορά το περιβάλλον, δημόσια υγεία, ασφάλεια τροφίμων και άλλα πράγματα που είναι σημαντικά προβλήματα ε, και είναι ζητήματα τα οποία δεν έχουν γεωγραφικό περιορισμό. Γιατί εδώ πέρα τα σύνορα δεν εκπληρώνουν πλήρως τον ε, ρόλο τους γιατί δεν χρησιμεύουν πολύ σε αυτή την περίπτωση. Επιπλέον, το δεύτερο το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι έχουμε 2.000 ευρωπαϊκά νομοθήματα τα οποία σήμερα ισχύουν για ζητήματα περιβάλλοντος, κλιματικής αλλαγής, δημόσιας υγείας, ασφάλειας τροφίμων και ισχύουν ε, και για το Ηνωμένο Βασίλειο και είναι σαφές ότι ένα Brexit θα έχει τεράστια επίδραση σε αυτά τα ζητήματα. Και επίσης, και αυτό είναι το τρίτο, είναι σαφές ότι αυτά τα 2.000 νομοθετήματα και οι ρήτρε ασφαλείας που έχουν δεν μπορούν απλά να εξαφανιστούν την ημέρα του Brexit. Βεβαίω πολλά από αυτά θα εξαρτηθούν από την μεταβατική περίοδο, γιατί μετά την αποχώρηση από το 2019 μέχρι το 2021 θα υπάρχει η μεταβατική περίοδος και εκεί πέρα θα ισχύουν πλήρως αυτά τα 2.000 νομοθήματα, δεν θα αλλάξει τίποτα. Αλλά μετά πρέπει να καθορίσουμε εντός αυτής της συμφωνίας μια συμφωνία σύνδεση δηλαδή με βάση το άρθρο 217, το πώς θα λειτουργεί. Και αν μου επιτρέπετε, θα έλεγα ότι θα έχουμε πέντε ερωτήματα κλειδιά που πρέπει να απαντηθούν και να απαντήσετε εσείς και να απαντήσουμε από κοινού στο ψήφισμά μας του Μαρτίου. Το πρώτο είναι πώς θα διασφαλίσουμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα διατηρήσει τις ίδιες παραγραφές περιβάλλοντος και τροφίμων, κάτι το οποίο έχει μεγάλη σημασία, ανδεδομένων και των μελλοντικών εμπορικών σχέσεων. Πώς θα γίνει αυτό. Δεύτερον, πώς θα εγγυηθούμε ότι οι μελλοντικές αποφάσεις του Ηνωμένου Βασιλείου ως ε, τρίτη χώρα δεν έχουν αρνητικό αποτέλεσμα στην υπόλοιπη Ευρώπη. Στην είναι η δεύτερη διασφάλιση και το δεύτερο πράγμα που ε, θα συζητούσα. Γιατί όταν βγουν θα είναι τρίτη χώρα. Εντάξει, στη μεταβατική περίοδο μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μεταβατική περίοδος, αλλά μετά θα πρέπει να φροντίσουμε οι αποφάσεις τους ε, να μην επηρεάζουν όλες τις πολιτικές μας. Το τρίτο ερώτημα νομίζω που θα πρέπει να απασχολεί στην Επιτροπή σας και να μας συμβουλεύσει είναι πώς να υπάρχει ταρχία πρόσβαση, κάτι που είναι σημαντικό για τους πολίτες, δηλαδή για τα ασφαλή φάρμακα για αυτούς που κατοικούν στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στην υπόλοιπη Ευρώπη των 27, διότι όταν θα είναι εκτός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, πώς θα μπορέσουμε να το εξασφαλίσουμε αυτό. Τέταρτον, Ελπίζω να το σκεφτείτε και αυτό για το ψήφισμα. Πώς θα δούμε το θέμα της αμοιβαία αναγνώρισης των σπουδών, των επαγγελματικών προσόντων, για αυτούς που θα δουλεύουν στον τομέα υγείας ιδιαίτερα. Και τέλος, πώς θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε της, την ανταλλαγή πληροφοριών ως προς την, ε, τις γνώσεις και τις πληροφορίες στον τομέα των γνώσεων και των πληροφοριών. Και τι μπορεί να γίνει ως προς την ασφάλεια τροφίμων σε μια χώρα που όταν αλλάξει η κυβέρνηση μπορεί να έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα νέο σοκ. Κύριε Στάς, μη γελάτε, ξέρετε ε, τι εννοούσα. Ήταν η ευκαιρία για το δικό σας κόμμα να μπει στην κυβέρνηση. Αυτά είναι τα πέντε κύρια ζητήματα, ίσως υπάρχουν και άλλα, αλλά σε αυτά θα πρέπει να δώσουμε μία απάντηση στο ψήφισμα όχι με μία εκατοντασέλιδη έκθεση, απλώς να γνωμοδοτήσουμε, να πούμε πώς πρέπει να έχουν και να λειτουργούν τα πράγματα. Και θα πρέπει να επηρεάσουμε και τις συναντήσεις έτσι ώστε να κινηθούμε προς τις κατευθυντήριες γραμμές που θα οριστούν. Χαίρομαι που με προσκαλέσατε για να μιλήσουμε για τις δικές σας υποδείξεις επί του θέματος. Ευχαριστούμε κύριε Φερχόφστατ. Επιστήσατε την προσοχή μας σε πολλά ζητήματα. Ορισμένα έχουν συζητηθεί στην Επιτροπή μας, δεν αποτελούν κάτι το καινούριο. Οι συνάδελφοι θα εκδηλώσουν μεγάλο ενδιαφέρον θα ήθελα όμως πριν δώσω το λόγο στους συναδέλφους να καλέσω τον κύριο Μπρόκ να σχολιάσει το θέμα. Θα ήθελα και εγώ να σας δώσω ορισμένες επιπρόσθετες πληροφορίες γιατί νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέχρι τώρα έχει ε, αντιδράσει στο θέμα σωστά. Και υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία. Σπάνια βλέπουμε τέτοια σύμπνοια σε τέτοια ζητήματα. Μπορεί ο συνάδελφος να μιλάει πιο κοντά στο μικρόφωνο. Θα κάνω ό,τι μπορώ παρόλο που λάμπω δια της παρουσίας μου. Το δεύτερο θέμα πολύ σημαντικό που ανέφερε ο Γκί είναι τα 60 σημεία. Τα 60 αυτά σημεία τα οποία μας απασχολούν ιδιαίτερα, δηλαδή να μην έχουμε ε, λανθασμένες προσδοκίες. Θα ήθελα λοιπόν να επικεντρωθείτε στα βασικά ουσιώδη ζητήματα. Ως προς τη μεταβατική περίοδο προχωρά όπως την ορίζουμε. Δεν θα πρέπει να υπάρξει πρόβλημα γιατί ισχύει το κοινοτικό και εκτιμένο. Έτσι προχωρούν τα πράγματα. Και θα πρέπει να ισχύσει το κοινοτικό και εκτιμένο και κατά την εφαρμογή της μεταβατικής περίοδου. Αυτό θα το ελέγξετε κι εσείς, αλλά δεν είναι μείζον ζήτημα. Στο μέλλον θα πρέπει να αναφερθούμε και στη Βόρειο Ιρλανδία. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι θα υπάρχει ένα αριθμιστικό πλαίσιο παρόμοιο μεταξύ αυτό της Ιρλανδίας με τη Βόρειο Ιρλανδία και θα πρέπει να επιλύσουμε θέματα περιβάλλοντος ασφάλειας και ούτω καθεξής γιατί θα υπάρχουν και πρακτικά προβλήματα. Και θα πρέπει να βασιστείτε στην πείρα σας. Ως προς την ε, περαιτέρω συμφωνία, πρόκειται για μια συμφωνία με μια τρίτη χώρα. Δεν πρόκειται για εξέλιξη της παρούσας κατάστασης. Είναι μια νέα συμφωνία με μία τρίτη χώρα, το οποίο σημαίνει διαπραγματεύσεις εξ αρχής, όπως κάναμε για παράδειγμα με ε, την εμπορική συμφωνία με τον ε, Καναδά. Θα πρέπει να δούμε πώς θα γίνουν επαναδιατυπώσεις των προδιαγραφών, έτσι ώστε να έχουμε μία ανοιχτή αγορά. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως ε, νομοθέτη θα αφορά ένα ρυθμιστικό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ κυβερνήσεων. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν θέλουν μία νορβηγική λύση οι Βρετανοί, γιατί αυτό σημαίνει θα πρέπει να καταβάλουν χρήματα, να ξαναδούμε εξ αρχής ε, την νομοθεσία και να πληρούν τους όρους των τεσσάρων ελευθεριών. Δηλαδή πρόκειται για μια ε, κλασική ε, συμφωνία, εμπορική συμφωνία πέρα από ζητήματα όπως το έρασμος και η ασφάλεια. Ως προς την εσωτερική αγορά και το περιβάλλον, ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο θα είναι η αλλιευτική συμφωνία. Το 93% των Βρετανών αλλιέων υπερψήφισαν το Brexit, αλλά τώρα θέλουν μεγαλύτερο μερίδιο της ευρωπαϊκής αγοράς. Μέχρι τώρα το 65% εξαγωγών πηγαίνει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους είπα ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ 93% και 65%. Δεν μπορώ να τα συμφιλιώσω αυτά τα δύο αριθμητικά στοιχεία. Θα πρέπει να δούμε και το σύστημα των ποσοστώσεων των υδάτων αλίευσης και νομίζω ότι είναι θέμα όχι μόνο της Επιτροπής Αλίας αλλά και της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Όλα τα άλλα ζητήματα αφορούν μία κλασική συμφωνία, εμπορική συμφωνία σε σχέση τώρα με, την, με τον τομέα της ε, δημόσιας υγείας αναφέρεται ότι το 70% των ε, φαρμακευτικών ε, σκευασμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο. Τώρα αυτό ίσως να αφορά τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων που τώρα θα φύγει από το Λονδίνο. Ναι, αλλά μιλάμε για τις έρευνες αυτές οι οποίες αυτή τη στιγμή γίνονται στο Λονδίνο. Θα παραμείνει αυτό το 70%. Δηλαδή, παίζει ρόλο ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, ναι ή όχι, γιατί έτσι κι αλλιώς θα μεταφερθεί από εκεί. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι το 70% των εξελίξεων στα φαρμακευτικά σκευάσματα προέρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό έχει να κάνει με τις φαρμακευτικές εταιρείες. Θα πρέπει να ελέγξουμε τα αριθμητικά στοιχεία και πάλι. Ναι, θα πρέπει να το αποσαφηνίσουμε, αλλά ίσως υπάρχει ένα θέμα κατανόησης και θα πρέπει να επανεξετάσουμε τα αριθμητικά στοιχεία. ως προς τα φαρμακευτικά σκευάσματα. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση μιας τρίτης ε, χώρας. Θα πρέπει να γίνουν έλεγχοι έτσι ώστε να ξέρουμε ότι οι δικές μας προδιαγραφές είναι οι ίδιες, ότι τηρούνται οι δικές μας προδιαγραφές. Τώρα, σε σχέση με την ε, διατροφική ασφάλεια και τα φαρμακευτικά σκευάσματα δεν θα πρέπει να υπάρχει αρνητική επίδραση έτσι ώστε να καταρρεύσει το σύστημα. Ίσως η Μεγάλη Βρετανία βρει μια ανοιχτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την καταβολή των εισφορών. Αναπροϊόν ή ανατομέα. Στον χρηματοπιστωτικό τομέα θα χρησιμοποιήσουν ε, το ίδιο επιχείρημα. Τα πράγματα έχουν τόσο καλά που θα πρέπει να συνεχίσουν ως έχουν. Γιατί Η Μεγάλη Βρετανία δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά χωρίς να καταβάλει το αντίτιμο. Δηλαδή, ε, αν δεν υπάρχει ελεύθερη κυκλοφορία εργασίας, κεφαλαίου κλπ. Θα πρέπει λοιπόν σε κάποιο σημείο να μην ξεχνάμε αυτά τα πολύ βασικά δεδομένα που έχουμε ε, στις κατευθυντήριες ε, γραμμές για το ψήφισμα και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μία ε, χώρα η οποία αποχωρεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να έχει τα ίδια δικαιώματα με μία χώρα η οποία παραμένει ή βρίσκεται εντός. Θα πρέπει να τιμήσουμε αυτή την ρίση γιατί διαφορετικά είναι σαν να στέλνουμε το μήνυμα ότι βγείτε, δεν έχετε να πληρώσετε τίποτα και προχωράμε όπως πριν. Αυτό λοιπόν είναι το σημείο εκκίνησης, ότι βγαίνετε και σας αντιμετωπίζουμε ως τρίτη χώρα και δεν μπορείτε αυτόματα να έχετε δικαιώματα χωρίς να τηρείτε υποχρεώσεις. Και όταν τα δούμε ανατομέα όλα αυτά. Ίσως φανεί ότι είμαστε αρκετά ανοιχτοί, αλλά το τελικό αποτέλεσμα θα είναι πολύ αρνητικό. Θα ήθελα λοιπόν να τηρηθεί αυτό το, αυτό το ρητό, δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχουν τα να υπάρχουν ίσα δικαιώματα. Δεν είναι τιμωρία, θα ήταν τιμωρία για τα κράτη μέλη τα οποία παραμένουν εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό το βλέπω και από το παράρτημά σας εδώ που διάβασα, να μην φανεί, να μην υπάρχει παρεξήγηση. Δηλαδή, ωραία. Όντως για κάποιους τομεί, όπω α πούμε η δημόσια υγεία τα πράγματα μπορεί να είναι λίγο πιο περίπλοκα αλλά εντάξει θα αφήσουμε και του συναδέλφου να σχολιάσουν όλα τα θέματα αυτά. Λοιπόν αρχίσουμε με του ε, συντονιστέ, Ο κύριο Λίζε πρώτα. Δυόμιση λεπτά παρακαλώ. Είναι ο κανένα για να μπορέσουμε να μιλήσουμε όλοι. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Κίφερ Χόφστατ, ευχαριστώ και τον Όλμαρ Μπρόκ. Η γενική γραμμή που μας παρουσίασαν και οι δύο Νομίζω ότι είναι απολύτως σωστή. Τη συμμερίζομαι απόλυτα. Τώρα για τη μεταβατική συμφωνία. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αποκλίνουμε από το κοινοτικό κεκτημένο, κυρίως για την υγεία, το περιβάλλον και την ασφάλεια τροφίμων. Και επίσης συμμερίζομαι αυτό που είπε και ο Γκί. Αν μιλούμε για πέραν του τέλους του 2020, μπορεί να είναι και καλύτερο τα πράγματα. Όσο πιο μεγάλη είναι η μεταβατική περίοδος, τόσο καλύτερα. Ίσως ε, ε, βρουν τα λογικά τους οι άνθρωποι να καταλάβουν ότι τελικά το Brexit είναι μάλλον κακή ιδέα. Δύο ερωτήματα έχω για το περιβάλλον. Έχω κάνει μια συζήτηση με την ε, χημική βιομηχανία της Γερμανίας, η οποία λέει ότι το πιο σημαντικό είναι να παραμείνει το REACH ως έχει να χρησιμοποιήσει δηλαδή το Ηνωμένο Βασίλειο το REACH, να συνεχίσει να το, να το χρησιμοποιεί. Αυτή είναι η άποψη της, γενικής, της χημικής βιομηχανίας και επίσης και στο Ηνωμένο Βασίλειο και ο υπουργό Περιβάλλοντος του Ηνωμένου Βασιλείου είπε ότι δεν θέλει λιγότερη προστασία περιβάλλοντος αλλά περισσότερη και έχω την υποψία ότι μάλλον ε, προσπαθεί να βρει ε, επιχειρήματα υπέρ του Brexit, όχι γιατί πραγματικά τα θέλει. Οπότε θα ήθελα παρακαλώ την ε, εκτίμηση των δύο συναδέλφων. Και μετά για την υγεία. Όντω είναι δύσκολο αυτό το 70% δεν το πιστεύω εγώ και θα ήθελα αν υπάρχουν περισσότερε πληροφορίε να μου τι δώσετε γιατί δεν νομίζω ότι είναι 70% τουλάχιστον από του δικού μου υπολογισμού. Ε, βιομηχανία, γιατροί, ασθενεί, και η Βρετανική κυβέρνηση μας τα λέει ότι για την υγεία θέλουμε να τα αφήσουμε όλα έτσι όπως είναι. Πριν το συζητήσουμε όμως αυτό, καλό θα ήταν να μας πούνε οι Βρετανοί τι ακριβώς θέλουν να κάνουν. Όταν έρχεται η Βρετανική κυβέρνηση και μας λέει ότι πρέπει να μείνουν τα πράγματα όσο έχουν, καταρχάς πρέπει να το πει ο υπουργό. Ψηφίσανε για τον Brexit, οπότε αυτό το θεωρούμε πλέον δεδομένο. Αν τώρα τα πράγματα αλλάξουν, εντάξει, να το συζητήσουμε. Αυτή τουλάχιστον είναι η δική μου εκτίμηση και νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε γενικότερα τα πράγματα και τις διασυνδέσεις, έτσι όπως μας παρουσίασε ο Έλμαρ Μπροκ. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, ο κύριος Ντάνς. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα. Πάντα με στεναχωρείτε όταν μιλάτε για το Ηνωμένο Βασίλειο ω τρίτη χώρα. Βεβαίω αυτό πρέπει να κάνετε, αλλά παρόλα αυτά με στεναχωρείτε. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν πολλοί που είναι αντίθετοι με τον Brexit, το ξέρετε αυτό και θα συνεχίσουν να το κάνουν. Πέραν αυτού, το Brexit συμβαίνει, εξελίσσεται και υπάρχουν πολλά που μα είπατε ότι είναι όντω πολύ σημαντικά. Για τη μετάβαση. Ναι, είναι πολύ σημαντικό να παραμείνει το status όσο έχει, κυρίω για δύο λόγου. Καταρχά, για να υπάρξει μια συνέχεια και μια ασφάλεια που χρειαζόμαστε και δεύτερον οι επιχειρήσεις λένε ότι δεν θέλουν δύο αλλαγέ, θέλουν μία. Οπότε νομίζω ότι αυτό που μας αναφέρατε είναι απολύτως λογικό. Όχι ότι αυτό δεν θα δημιουργήσει βεβαίω πολιτική καταιγίδα ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο, φυσικά. Τώρα, για τα διάφορα πρότυπα. Είπανε πολλοί ότι το Brexit είναι ευκαιρία να ε, επιδεινώσουμε τα πράγματα, να φύγουν, να, να καταργήσουμε όλες τις ασφάλειες που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή μάλιστα είναι η φιλοδοξία πολλών του κυρίου Φάραντς και άλλων όσων έχουν δηλώσει παρόμοια πράγματα. Στο ψήφισμα θα είναι σαφές ότι για το μέλλον και για τις εμπορικέ μας σχέσεις στο μέλλον οποιαδήποτε συμφωνία, ελεύθερο εμπορίο ή οτιδήποτε είδους είναι θα υπάρχει σαφής αναφορά στις, ε, στο ότι η νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος είναι σε ισχύ. Γιατί για την Ευρωπαϊκή Ένωση προφανώς αυτό είναι το ελάχιστο. Οι χώρες μπορούν βεβαίως να ενισχύσουν αυτούς τους κανόνες. Αλλά αυτό θα ήταν πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η ε, ρήτρα. Και επίσης ότι το, ε, αν φύγουμε από το ε, δικαστήριο σημαίνει ότι οι, οι δυνατότητες επιβολής από την πλευρά της κυβέρνησης τίθεται ένα αμφιβόλο αλλά και, τα, και η δυνατότητα των πολιτών να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους τίθεται ένα αμφιβόλο. Τι μπορούμε λοιπόν να πούμε ε, μέσα σε αυτό το ψήφισμα που να κάνει ρητή αναφορά και μνήα στη δυνατότητα να, να εφαρμόσουν νομικώ όλα αυτά τα πρότυπα. Και ένα τρίτο σημείο. Πρόσβαση στα φάρμακα. Πρέπει να είναι προτεραιότητα στη δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων. Να εξασφαλίσουμε ότι η προσφορά ε, φαρμάκων στους ε, ασθενείς θα διασφαλίζεται και να έχουμε διαπραγματευτικές εντολές έτσι ώστε να υπάρξει ποιότητα και προσφορά φαρμάκων. Αυτό θα πρέπει να είναι ένα βασικό στόχο μα. Καταλαβαίνω ότι ο Έλμαρ Μπροκ λέει ότι δεν μπορείτε να μα δώσετε λεπτομέρειε, αλλά πρέπει να υπάρξει σαφή υποχρέωση στο ψήφισμα ω προ αυτό, γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Η κυρία Γκέρλινγκ, ευχαριστώ. Το ερώτημά μου είναι παρόμοιο με αυτό του ΣΕΜ. Θέλω κι εγώ λίγο να καταλάβω πώ θα είναι οι ε, μελλοντικέ εμπορικέ σχέσεις μας με το Ηνωμένο Βασίλειο σε σχέση με τις, υποχρεω... για το περιβάλλον. Γιατί σωστά είπατε ότι αυτά που υπάρχουν τώρα είναι το ελάχιστο για να είναι κανεί μέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης οπότε και τη ενιαία αγορά. θα πρέπει να υπάρχει και κάποιο ε, περιβαλλοντική πτυχή. Αυτό που με ανησυχεί εντωμεταξύ είναι ότι οι περιβαλλοντικέ πτυχέ δεν έρχονται ποτέ στο προσκήνιο. Ε, Τι συζητούμε μεν γιατί ίσω είναι ένα θέμα τη μόδα, αλλά δεν νομίζω ότι ποτέ θα αποτελέσει το σημείο που θα, που θα ε, καταστρέψει μια συμφωνία. Οπότε παρακαλώ να το θεωρήσουμε πιο σημαντικό θέμα. Και επίσης, αυτό που είπε ο κύριο Μπροκ για τις λεπτομέρειες. Ε, προφανώς δεν μπορείτε να μας πείτε λεπτομέρειες. Το θέμα είναι να καθορίσουμε κάποιες αρχές. Δεύτερον, όταν μιλούμε για τη μεταβατική περίοδο, δεν είναι σαφές για μένα τι θα πει αυτό. Είναι σαν να λέμε ότι παρατείνεται το άρθρο 50 και οι σχετικές διαπραγματεύσεις. Γιατί θα υπάρχουν τόσα πολλά που πρέπει να συμφωνηθούν κατά τη διάρκεια τη μεταβατική περίοδου. Και σίγουρα τα περισσότερα από τα περιβαλλοντικά σημεία εκεί θα έχουν διαπραγμάτευση. Οπότε αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι αφήνουμε μια συμφωνία να εδρεωθεί. Ε, δεν νομίζω ωστόσο ότι θα υπάρχουν λεπτομερεί συμφωνίε για τούτη την μεταβατική περίοδο. Και ένα ερώτημα για το Κοινοβούλιο. Εγώ ω μέλο του, του Βρετανικού Κοινοβουλίου ή εκπρόσωπο του Βρετανικού Κοινοβουλίου δεν θα είμαι μέλο του Ευρωπαϊκού από τα μέσα του επόμενου έτου, αλλά το Κοινοβούλιο θα εξακολουθήσει να έχει ε, δυνατότητα έκφραση θέση για τη συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, χωρί όμω τη συμβολή των Βρετανών ε, Ευρωβουλευτών. Εσεί πώ το βλέπετε αυτό να εξελίσσεται και πώ θα λειτουργήσει η δική σα η ομάδα, α πούμε, κατά τη διάρκεια τη μεταβατική περίοδου. Και επίση θα υπάρχει κάποια συμβολή από κάποια βρετανική φωνή σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκερμπράντη. Θα μιλήσω εγώ εκ μέρους του Άλντε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε για την παρουσίασή σας. Όπως και ο Σεμπ και η Τζούλη όταν αναφέρεστε σε εμά ω τρίτη χώρα είναι ε, οδυνηρό και να υπάρχουν άνθρωποι που ακόμη αντιτίθενται σε αυτό. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πάνω από 40 χρόνια μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε υιοθετήσει ένα μεγάλο αριθμό ε, περιβαλλοντική νομοθεσία και περιβαλλοντικών συμφωνιών και μάλιστα είμαστε μέρος της προσπάθειας που γίνεται να προωθηθούν οι ε, προσπάθειες για να επιτύχουμε τους στόχους. Είμαστε μέρος του Συμφωνίας των, ε, των Παρισίων για την προστασία της άγριας ζωής, για τη μείωση των εκπομπών, ε, προστασία επίσης για την οδηγία για τους βιοτόπους κτλ δεδομένης και της ε, υφή των ε, περιβαλλοντικών προβλημάτων. Θα ήταν καταστροφικά αν το Ηνωμένο Βασίλειο απλώς αποχωρούσε από τις υποχρεώσεις του για την επιβολή των περιβαλλοντικών προτύπων όπως συμβαίνει στο υπόλοιπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χαίρομαι που το αναφέρετε. Η κυρία Μέη και ο Υπουργό ε, Περιβάλλοντος έκαναν ένα σχέδιο 25 ετές για το περιβάλλον αλλά σήμερα ακούμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο καθυστερεί και στυλώνει τα πόδια στο Συμβούλιο για τον στόχο του 65% των λιμάτων μέχρι το 2035 για τα απόβλητα. ακόμα λοιπόν και αν στην αρχή θέλαμε να προωθήσουμε τις προσπάθειες αυτές, βλέπουμε ότι τώρα τα πράγματα δεν είναι έτσι. Και μάλιστα μπορούν να, τώρα θέλουν να καταρρύψουν και 40 χρόνια προσπαθειών για την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων. Δεν είμαστε τρίτη χώρα που πρέπει να αυξήσει τα πρότυπά τη. Ήδη σε μεγάλο βαθμό είμαστε συμμορφούμενοι με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και αν δεν το κάνουμε αυτό υπάρχει κάποια κύρωση. Αλλά το μάντρα του δημοψηφίσματος ήταν ότι πρέπει να πάρουμε πίσω τον έλεγχο. Οπότε αν είμαστε τώρα στο, ήδη στο επίπεδο αυτό, το να πάρουμε πίσω τον έλεγχο σημαίνει ότι θα μειώσουμε τα πρότυπα που έχουμε και το πώς θα εφαρμοστούν αυτά από την πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να το δούμε. Αυτή τη στιγμή έχει αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αλλά οι ποινέ ποιε θα είναι και πώς θα επηρεαστεί αυτό από την, πώς θα επηρεαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση από αυτές. Όχι μόνο για τα φάρμακα. Έχουμε να μιλήσουμε για εμπόριο, πούμε, ε, προϊόντων άγρια ζωή. Ε, παράνομο προφανώ. Ε, δεν μιλάμε δηλαδή μόνο για το ε, περιβάλλον, μιλάμε και για άλλους ε, τομείς. Έτσι ώστε να καταλήξουμε τελικώ σε μια διεθνή συμφωνία με όλες τις δικλείδες ασφαλείας που έχουν οι διεθνείς συμφωνίες απανταχού της γης. Πρόσβαση στα φάρμακα επίσης. Είναι, δεν είναι μονόδρομος. Μην το ξεχνάτε αυτό. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ο κύριος Φλάνεγκαν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε να σας κάνουμε ερωτήσεις. Είστε βασικά, ήσασταν ο διαπραγματευτής μας ε, για το Brexit. Ε, εγώ όταν εξελέγη μου είπα να εκπροσωπήσω τις απόψεις των ψηφοφόρων μου και τώρα τελικά εσείς θα τις εκπροσωπήσετε, τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δηλαδή, επί του Brexit ε, κατά την απόψή μου. Είστε εδώ, κάνετε ήδη την δουλειά, εντάξει δεν είστε ο ιδεώδης δεδομένων των απόψεών σας για αυτό το οποίο θέτε δηλαδή οι Ηνωμένε Πολιτείε της Ευρώπης και το Ηνωμένο Βασίλειο έφυγε ακριβώς γιατί υπήρχε αυτή η φούρια για περισσότερη ολοκλήρωση και εσείς είστε σύμβολο αυτής της ε, διαδικασίας και είχατε περιγράψει το Ηνωμένο Βασίλειο ως νάνο αν φύγει. Η ανησυχία μου και η ερώτηση που έχω είναι θα αποδειχτείτε σωστός ε, κάνοντας την ε, Αγγλία έναν νάνο, κάτι το οποίο θα μας δημιουργήσει τρομερά προβλήματα στην Ιρλανδία, καθώς εξαρτώμεθα. Ε, έχετε φύγει από αυτή την ιδέα ότι πρέπει να είναι νάνος το Ηνωμένο Βασίλειο όταν φύγει επίσης. Ε, τι σχέση είναι αυτή όταν λέτε σε κάποιον ότι δεν πρέπει να σας αφήσει γιατί θα γίνει νάνος, είναι εγγύηση ότι την άλλη μέρα θα φύγει. Και πρέπει να βασιζόμαστε σε εσά όμως λέτε ότι συνεισφέρουν και οι άλλες επιτροπές στην δική σας διαπραγματική εντολή. Φανταστικό αυτό και στην Άγκρη το ίδιο έγινε. Συζητείτε το να προσκαλέσετε εαυτόν ε, μαζί με τον κύριο Μπαρνιέ. Το θέμα είναι τι μορφή θα έχει αυτή η συνεργασία. Λέτε ότι το ψήφισμα θα έρθει στις Επιτροπές προσέγγιση αφού συνταχθεί. Δεν θα ήταν πιο λογικό να μας μιλήσετε εκ των προτέρων, να έχουμε κάποια ε, επίσημη δομή. Ξέρω πως ο χρόνος ε, θα είναι πρόκληση. Και δύο ακόμα ερωτήσεις. Πού νομίζετε θα πρέπει να είναι το σύνορο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου. Και βεβαίως μας απασχολούν πολύ το αλλά τι θα γίνει με την αλληλεία τώρα που δεν θα είναι πλέον η ε, δεν θα έχουν οι ευρωπαϊκοί στόλοι την δυνατότητα να αλλιεύουν στα βρετανικά ύδατα. Θεωρείτε ότι θα έρθουν στα Ελλανδικά. Καλή τύχη σας εύχομαι. Δεν συμφωνούμε στα πάντα, αλλά ε, πρέπει να κάνετε καλή δουλειά. Ευχαριστώ κύριο Τέιλορ. Ναι, ναι, εσείς, ναι. Ναι, ναι, συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίασή σας και την ευκαιρία που μας δίνετε να πούμε κάποια πράγματα. Θα επικεντρωθώ σε ένα πράγμα. Συμφωνώ με την άποψη των περί κομμάτων εδώ, αλλά αυτό το οποίο θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι το εξή. η ενημέρωση την οποία στείλατε μιλούσε για το περιβαλλοντικό και εκτιμένο. Αλλά εμένα με ενδιαφέρει επίσης ε, και η ευζοία των ζώων που δεν αναφέρεται εδώ, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό και δεν πρέπει να το παίρνουμε ελαφρά, ειδικά όταν μιλάμε για παραγωγικά ζώα, για ζώα συντροφιάς και για πειραματόζωα εργαστηρίου. Έχουμε διάφορα νομοθετήματα που αφορούν αυτά τα ζητήματα που επηρεάζουν το εμπόριο που θα πρέπει να διασφαλιστεί ε, για το όφελος της Ευρώπης. Γιατί ποιος ξέρει τι θα γίνει μετά το Brexit. Εάν η Βρετανική κυβέρνηση αποφασίσει ότι θέλει να έχει υψηλότερες ε, προδιαγραφές, παραδείγματο χάρη, για το σπιτικό βοδινό ή για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Εάν θέλουμε λοιπόν να μειώσουμε κάτι τέτοιο, θα πρέπει να, τέτοιες προδιαγραφές θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα αναφέρουμε συγκεκριμένα την ευζοία των ζωών στο ψήσιμο. Ευχαριστώ και θα ήθελα να ακούσω την απάντηση. Thank you. Now, Reed. Ευχαριστώ. Κύριε Ρο, Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σε αντίθεση με πολλούς συναδελφούς, εγώ θεωρώ το Brexit θα είναι ευκαιρία για την Βρετανία και Βεβαίω, ε, διάφορα νομοθετήματα της Ένωση έχουν προκαλέσει προβλήματα, μεταξύ των οποίων η γεωργική πολιτική. Η δημιουργία αυτών των τεράστιων ε, αγροκτημάτων ε, έχει οδηγήσει στην καταστροφή των παραδοσιακών φραχτών στη Βρετανία γη στην δική μου την περιοχή φύτευαν ε, σε μέρη τα οποία έπρεπε να είχαν καθίσει σε αγρανάπαυση και ε, μετά έσπερναν στον ε, κάμπο. Ένας δε μελισσοκόμος φίλος μου διαπίστωσε ότι οι μέλισσες πεινούσαν γιατί τα τεράστια αυτά τα χωράφια είχαν μόνο δημητριακά και δεν υπήρχε τίποτα ε, με γύρι για τις μέλισσες. Κάτι άλλο αφορά τις ποσοστώσεις ε, γάλακτος ε, και τα αγροκτήματα πλέον δεν, οι εκμεταλλεύσεις δεν έχουν αγελάδες. Και εγώ θεωρώ λοιπόν ότι έχουμε μια ευκαιρία. Ο Υπουργό ο κύριος Γκόβ είπε ότι θα εξετάσει και τα ζητήματα των άγριων φυτών και των βοσκοτόπων. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι μια ευκαιρία να τα πάμε καλύτερα και προφανώς ε, θέλουμε να εμπορευτούμε. Είμαστε φίλοι με τους γείτονές μας αλλά θέλουμε να έχουμε και την ευκαιρία να γράφουμε μόνοι μας τους νόμους μας και ελπίζω να καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία χωρίς να μας λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση το τι πρέπει να κάνουμε σε δέκα χρόνια από σήμερα. Ωραία. Κυρία Μελά. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ενημερώσατε για το στάδιο των διαπραγματεύσεων. Κατέγραψα τα πέντε ερωτήματα επί των οποίων θα επιμείνετε. Το πρώτο σημείο αφορά τις, ε, τα ίδια πρότυπα που ισχύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα γι' αυτά τα πρότυπα αποχώρησαν οι Βρετανοί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος ε, Μπρόκ μίλησε για τις αξιώσεις των Βρετανών. Νομίζω ότι όλοι έχουν έχουμε ε, προσδοκίες, αλλά προσδοκίες προς τα κάτω και το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να λάβει υπόψη τις ε, συνέπειες ε, της επιλογής του. Ο κύριος Φλάναγκαλ μίλησε για τα σύνορα που θα πρέπει να ισχύσουν για την Ιρλανδία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στο καλέ έχουμε χιλιάδες μετανάστες Έχουμε καταβλισμούς, άλλοι οι ε, πολλοί από αυτούς τους μετανάστες ζητούν άσυλο και 90% βεβαίως ε, βλέπουν την αίτησή τους να απορρίπτεται φεύγοντας αλλά ξαναγυρνώντας στο καλέ για τα ίδια διαβήματα. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε σαφείς για το πού ε, βρίσκονται τα σύνορά μας και έχουμε πολύ υψηλές προσδοκίες από εσάς. Η κυρία Μακίνες. Ευχαριστώ και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Φερχόφστατ και Μπροκ για την παρουσίαση τους και γιατί μας υπέβαλαν πέντε ερωτήσεις για το πώς. Και θα ξέρουμε την απάντηση μόνο όταν μάθουμε τι θα αποφασίσει το Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, σε σχέση με την ασφάλεια για τα φαρμακευτικά σκευάσματα ή για τους ασθενείς ως προς την πρόσβαση στα φάρμακα υπάρχουν 45 εκατομμύρια σκευάσματα που ε, προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο και φτάνουν στο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ 37 είναι ο αντίστοιχος αριθμός προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν ξέρω τι νομίζετε ότι θέλει το Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί από όσο ακούω το Ηνωμένο Βασίλειο θέλει να παραμείνει κοντά, αλλά δεν ξέρουμε πώς. Ως ως προς τη διασυνοριακή μετακίνηση και το σύστημα υγείας έχουμε μια πολύ καλή διασυνοριακή ε, ανταλλαγή απόψεων για το σύστημα υγείας. Το έχω συζητήσει με τους Ιρλανδούς, αλλά θα ήθελα να τονίσω ότι υπάρχουν πραγματικά θέματα ασφάλειας των ασθενών εάν αποκλίνουμε από το σύστημα όπως είχε ε, συσταθεί και από όσο μας είπαν οι ασθενείς θέλουν να παραμείνουν στο ε, παρόν καθεστώς. Ε, ξέρουμε ότι και η Νορβηγία το θέλει, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι θέλει το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό αφορά και την προστασία του περιβάλλοντος και την τροφική ασφάλεια. Το θέμα είναι ανησυχητικό, γιατί αν το Ηνωμένο Βασίλειο φτάσει σε εμπορικές συμφωνίες με τρίτες χώρες, θα πρέπει να δούμε πώς θα αλλάξουν οι προδιαγραφές της για την ασφάλεια των τροφίμων. Αυτή τη στιγμή διαπραγματευόμαστε μέσα στα πλαίσια ενός χάσματος, γιατί δεν ξέρουμε επακριβώς τι θέλει το Ηνωμένο Βασίλειο και δεν ξέρουμε πώς να προστατεύσουμε τους πολίτες και τις αγορές μας. Λάινεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όταν βγει από την ε, εσωτερική αγορά του Ηνωμένο Βασίλειο, νομίζω ότι πρέπει να φοβόμαστε ότι θα φτάσουμε ή θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε διαφορετικά πρότυπα για την ασφάλεια των τροφίμων, για το περιβάλλον και για την υγεία. Πολλές φορές έχει ανακοινώσει το Ηνωμένο Βασίλειο ότι θέλει διαφορετικά πρότυπα. Η Τερέζα Μέη ούτε καν για τους, ε, με τους στόχους μας για, το, για τα πλαστικά δεν συμφωνεί. Οπότε δεν νομίζω τα πράγματα θα είναι καλύτερα, μάλλον χειρότερα θα είναι. Όπως και σε άλλες τέτοιες ε, συνθήκες ε, προσπαθούμε μέσω της ε, Ρυθμιστικής Επιτροπής να διατηρήσουμε έναν έλεγχο στα πράγματα, αλλά εδώ πρέπει να πω ότι είμαστε 27 χώρες και το Ηνωμένο Βασιλείο είναι μία. Δεν γίνεται να, ο Μουτζούρης να κανονίζει πώς θα παιχτεί το παιχνίδι. Δεν μπορεί να μας τραβήξει προς τα κάτω το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό θα πρέπει να του το πούμε ξεκάθαρα. Ένα θέμα ήθελα εγώ να θίξω. Νομίζω ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποχωρήσει και από τη συνθήκη Ευρατών και από εκεί απορρέουν πολλά ερωτήματα. Γιατί έχουν πυρηνικό υλικό, έχουν πρότυπα για, πρότυπα για τους πυρηνικούς σταθμούς, έχουν πυρηνικά απόβλητα, διασυνοριακές πληροφορίες για ατυχήματα. Υπάρχουν λοιπόν πολλά ερωτήματα που προκύπτουν αν όντως αναχωρήσουν και από την συνθήκη Ευρατών. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λόρενς. Ευχαριστώ. Ακούγοντάς σας, νομίζω ότι ε, περιμένετε κι εσείς να αλλάξουν τα πρότυπα. Αλλά αν αλλάξουν τα πρότυπα, οι 27 χώρες πόσο προετοιμασμένες είναι να δεχτούν ή να εξετάσουν τα νέα πρότυπα του Ηνωμένου Βασίλειου. Μιλάμε για χρήση υλικών, για διάφορα θέματα. Πόσο μπορούμε να ελέγξουμε εμείς ή τα κράτη-μέλη μια νέα συμφωνία με μια τρίτη πλέον χώρα. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ πρόεδρε. Κατανοώ ότι υπάρχουν ανησυχίες στον τομέα της υγείας όπως και άλλα θέματα που αφορούν το Brexit. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχουμε εμείς μεγάλο πρόβλημα από όσο ακούμε τους διαφόρους εκπροσώπους το Ηνωμένο Βασίλειο, το πρόβλημα αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο και όχι εμάς. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα απομακρυνθεί από τα δικά μας πρότυπα υγείας. Γι' αυτό νομίζω ότι εκείνοι απομακρύνονται και θα είναι δύσκολο να φτάσουμε σε μία συμφωνία εάν απομακρυνθούν από τα δικά μας πρότυπα. Εάν μιλάμε για το προσωπικό, υγείας πρόκειται για 144.000 που δεν έχουν την ε, βρετανική υπηκότητα, δηλαδή 14% του συνολικού προσωπικού υγείας. Από ό,τι ξέρω δεν υπάρχει καμία εγγύηση για αυτούς τους επαγγελματίες οι οποίοι ενδεχομένως θα πρέπει να επιστρέψουν στις χώρες τους. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να διευκολύνουμε το θέμα αυτό των επαγγελματικών προσόντων και της αναγνώρισης τους ως προς το... την έρευνα στον ιατρικό τομέα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ποιες θα είναι οι συνέπειες και νομίζω ότι η αριστεία αυτή που υπάρχει στο Ηνωμένο Βασίλειο αφορά και το δικό μας ε, πρόγραμμα. Εάν πρόκειται για ένα 70% θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Σε θέματα έρευνας θα πρέπει να δούμε ότι υπάρχει μια προστιθέμενη αξία την οποία ίσως χάσουμε. Μας ενδιαφέρει λοιπόν να υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση και το σημείο εκκίνησης θα πρέπει να είναι τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούμε να τα χάσουμε ούτε στον τομέα της υγείας. Θα πρέπει να διενεργηθούν μελέτες για, νομίζω, για να δούμε, όπως νομίζω εγώ, πώς θα κινηθούμε στο μέλλον. Ωραία, έτσι συνεισέφεραν όλα τα μέλη. Ο κύριος Μπροκ, καταρχήν, να μας πείτε πώς βλέπετε τα πράγματα. Ευχαριστώ να αναφερθώ σε κάποια πράγματα. Δεν μπορώ να απαντήσω σε όλα και Ζητώ συγγνώμη γιατί έχω να βγάλω ομιλία στην περιφέρειά μου. Ναι, ναι, το, το σημαντικότερο, το σημαντικότερο είναι αυτό. Λοιπόν, να απαντήσω στα γερμανικά. Θεωρώ πως η μεταβατική ρύθμιση και γενικεύω τώρα λίγο σημαίνει όπως το αντιλαμβανόμαστε εμείς ότι παραμένουν οι προδιαγραφές που ισχύουν σήμερα. Κατά βάση αυτό ισχύει. Και κατόπιν, εάν υπάρξει μια επιτυχής διαμόρφωση, θα έχουμε μια συμφωνία την οποία θα διαπραγματευτούμε με μια τρίτη χώρα. Δεν θα έχουμε συνέχεια των υφισταμένων. Θα έχουμε κάτι το τελείως καινούριο. Γιατί ακούω καμιά φορά πράγματα από το Λονδίνο και εδώ μέσα. Και έχω την εντύπωση ότι εξηγούν οι οπαδοί του Brexit ότι τα πράγματα θα παραμείνουν όσο έχουν. Οι δε ημερίδε ημερίδες ε, μοιάζουν σαν να είναι αίτηση για ένταξη χωρίς τις υποχρεώσεις. Ε, δηλαδή την ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων, το ΔΕΚ και τα λεφτά. Και έχω ζήσει κάποια τέτοια παραδείγματα. Ή, ή τουλάχιστον εγώ έτσι τα κατάλαβα κάποια επιχειρήματα στον τομέα των φαρμακευτικών προϊόντων προσπαθούν να μας το εξηγήσουν. Είναι το ίδιο που ακούμε με τους Γερμανούς. Πώς μπορούμε να τους αντιμετωπίζουμε έτσι όταν πουλάει τόσα πολλά αυτοκίνητα ή BMW στην Αγγλία. Όχι, δεν πάει έτσι. Είναι συμφωνία με μια τρίτη χώρα. Όποιος έλαβε την απόφαση πρέπει να υποστεί και τις συνέπειες. Ε, πρέπει να γίνουν τα πράγματα ξεκάθαρα και υπ' αυτές τις συνθήκες να βρούμε μια επικοδομητική λύση. Και νομίζω ότι ε, έτσι θα γίνει. Η Βρετανία απορρίπτει την λύση της ε, Νορβηγίας γιατί δεν θέλει τις σχετικές υποχρεώσεις και θέλει μια συμφωνία ελευθερού εμπορίου. Αλλά μετά λέει η συμφωνία ελευθερού εμπορίου συν συν συν ουσιαστικά την εσωτερική αγορά. Και νομίζω ότι αν δούμε την συνολική εικόνα πρέπει να έχουμε κατά νου πως ε, στις λεπτομερίες δεν θα μπορέσουμε μετά να οδηγηθούμε σε μια πλήρη συμμετοχή της Μεγάλης Βρετανίας. Δεύτερον, μπορούμε να είμαστε πιο γενναιόδοροι σε μια εμπορική συμφωνία και αυτό είναι προς το αμοιβαίο συμφέρον μας. Αρκεί να τηρεί τις προδιαγραφές της Μεγάλη Βρετανία. Και αναφέρθηκε το ζήτημα της ε, Ρυθμιστικής Επιτροπής. Το έχουμε συζητήσει και στο πλαίσιο της TTIP. Εγώ είμαι κατά μια τέτοιας επιτροπής η οποία θα, καθαρί, θα καθορίζει κανόνες για εμάς και στην οποία δεν θα συμμετέχει το Κοινοβούλιο. Οποιαδήποτε ρύθμιση θα πρέπει να σέβεται την κυριαρχία του Κοινοβουλίου και να μην τα κανονίζουν υπάλληλοι μεταξύ Λονδίνου και Βρυξελών. Ξεκάθαρα. Και όταν η Μεγάλη Βρετανία λέει ότι εμείς θέλουμε την αυτονομία μας, δεν έχω καταφέρει να αντιληφθώ τι ακριβώς εννοούν. Δηλαδή θέλουν ε, να, υπάρχει ένα εμπόριο χωρίς δυσκολίες. Ελπίζω να με βοηθήσουν να το αντιληφθώ τους επόμενους μήνες οι βρετανικές προτάσεις, γιατί δεν έχω καταλάβει τι θένε. Και δεν πρόκειται βεβαίως να περάσουμε σε μια λανθασμένη τέτοια πορεία. Και νομίζω ότι και αυτά τα οποία ε, είπε ο Πίτερ για τον Μάικλ Γκόβ. Ο Μάικλ Γκόβ που ήταν ε, εκ των φανατικότερων υπέρ του Brexit. Ο οποίος εξήγησε ότι θέλει να φύγει από αυτή την ευρωπαϊκή γραφειοκρατία. Και βεβαίω ε, από τους ίδιους ανθρώπους που λένε ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μεγάλο κομμάτι αυτής της γραφειοκρατίας και τώρα λένε να τηρηθούν κάποιες ε, Πάλι δεν καταλαβαίνω το τι γίνεται. Τώρα το τι είναι προπαγάνδα και το τι όχι με αυτά τα οποία άκουσα εδώ πέρα για χωράφια και αγράβα αναπαύσεις δεν θα το σχολιάσω. Επίσης πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι στην ποιότητα των ε, προϊόντων θα εξετάζουμε. Την σχέση μας με τη Μεγάλη Βρετανία όπως κάνουμε με οποιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα. Τώρα, κάποιος είπε ότι θέλει η Μεγάλη Βρετανία να είναι μέλος στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων. Εντάξει, μπορεί να πληρώνει αν θέλει τη συμμετοχή, αλλά δεν θα συμμετέχει στη διοίκηση. Το ίδιο στη Europol. Χωρίς να είναι μέλος της διοίκησης, θα πληρώνει λεφτά. Άμα θέλει έτσι, είναι. Αλλιώς δεν έχει. Ε, είχα και μια συνάντηση με τον Νορβηγό πρέσβη και πληρώνουν οι άνθρωποι στο Εράσμους ή στο Horizon ακριβώς αναλογικά, αυτό που τους αναλογεί, ε, σύμφωνα με το ΑΕΠ, σαν να ήταν κράτος μέλος. Αλλά αν έχουμε κάποιες ε, αποκεντρωμένες υπηρεσίες και διαλέγουν τις υπηρεσίες που τους αρέσουν επειδή έχουν ένα πλέον πρέπει να δούμε το γενικότερο ερώτημα θεωρώ ότι στον τομέα της έρευνας και στα φάρμακα θα πρέπει να διατηρηθεί η συνεργασία και πανεπιστήμια και εταιρείε. Γιατί και η Μεγάλη Βρετανία προφανώς ε, μόνη της δεν έχει την κρίσιμη μάζα να είναι επιτυχημένη παγκοσμίω, αλλά από κοινού με εμάς θα μπορεί. Αλλά ταυτόχρονα το να πηγαίνουν οι 20-25% των κονδυλίων του Horizon στη Μεγάλη Βρετανία νομίζω δεν θα είναι αυτονόητο, θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης. το 1 τέταρτο των κονδυλίων για έρευνα του Horizon πηγαίνει στη Βρετανία. Και πρέπει να το σκεφτούν αυτό και οι του Brexit, το πώς θα το λύσουμε. Αυτά είναι οι πικρές αλήθειες ε, που έχουμε μπροστά μας. Κύριε Φλάναγκαν, η πολιτική σας ε, ομάδα είναι στο κατευθυντήρια επιτροπή του Brexit. Εκεί πέρα αποκαλύπτονται τα πάντα. Δεν κρύβουμε κάτι από την ομάδα σας. Και νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε μια καλή συνεργασία. Και να δούμε και τα ερωτήματα του κυρίου Τέιλορ τώρα με την ψωγεία των ζώων. Μα αυτό είναι κομμάτι των ευρωπαϊκών προδιαγραφών και για περιβαλλοντικούς λόγους και για λόγους ασφαλείας τροφίμων. Και ισχύει όπως όλες οι άλλες προδιαγραφές. Αν δεν πληρούν αυτούς τους όρους της ευσοίας ε, των ζώων υπάρχει πρόβλημα. Οπότε, θεωρώ, αυτό, λοιπόν, ο Καρλ Χάιντς ανέφερε κάτι μαζί με τον Πέτρε Λίζεκο. πρέπει να, για τις προδιαγραφές, σα δούμε το τι σημαίνει παραδείγματο χάρη η εφαρμογή του REACH για να το έχουμε ως υπόδειγμα συνεργασίας και του πώς μπορούμε να αναπτύξουμε προδιαγραφές προς το κοινό συμφέρον μας. Αλλά σας παρακαλώ. Να ε, λέμε ότι θα έχουμε συμφωνία μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να το ξεκαθαρίσουμε. Ο Γιολάινεν ανέφερε επίσης κάτι σημαντικό, η Ευρατόμ. Όχι μόνο στο θέμα του σχάσιμου υλικού, αλλά και στο θέμα του ελέγχου ασφαλείας. Ε, ένα άλλο το πρόβλημα μεγάλης σημασίας. Οπωσδήποτε θα αποτελέσει ξεχωριστό κεφάλαιο στις ε, διαπραγματεύσεις το τι σημαίνει η αποχώρηση από την Ευρατόμα από πλευράς οικονομικής, περιβαλλοντικής, ασφαλείας. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να πάμε στις ε, λεπτομερείς διαπραγματεύσεις. Τώρα εμείς καθορίζουμε τις κατευθυντήριες γραμμές ε, για τη δεύτερη φάση. Έχουμε λοιπόν την συμφωνία αποχώρησης που πρέπει να τεθεί εν μέχρι τον Μάρτιο, μετά θα έχουμε ταυτόχρονα θα έχουμε τις μεταβατικές ρυθμίσεις για να μην έχουμε την επόμενη μέρα κατάρρευση και να έχουμε δύο χρόνια να ε, καταλήξουμε σε μια λογική συμφωνία. Και ε, Νομίζω ότι το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να δούμε από κοινού ε, το ότι ε, τον, ε, το τέλος Μαρτίου 2019 η Μεγάλη Βρετανία είναι τρίτη χώρα. Και υπάρχει αυτό το πλαίσιο λαμβάνουν χώρα οι διαπραγματεύσεις καθαρά και μιλημένα για να μην υπάρχουν εδώ πέρα ψευδεστήσεις και να μην ακούμε τέτοιες ε, παρατηρήσεις ε, τώρα περί συνόρων ε, μετανάστευσης και Μεγάλης Βρετανίας. Και, γιατί στο δημοψήφισμα έλεγαν ότι είναι υπεύθυνη η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μετανάστευση στη Μεγάλη Βρετανία. ανακάτευαν δηλαδή την ελεύθερη μετακίνηση των Πολωνών με τους πρόσφυγες ε, από το Σύρια και το Ιράκ. Η Γαλλία ε, καταβάλει μεγάλες προσπάθειες στο Καλέ. Η Μεγάλη Βρετανία δεν είναι στο Σέγγεν και πάντα έλεγχε τα εξωτερικά της σύνορα. Δεν έχει να αποκαταστήσει τίποτα γιατί δεν το είχε ποτέ παραδώσει. Η Γαλλία προστάτευσε την Μεγάλη Βρετανία και δεν άφηνε, το, δεν άφηνε τον κόσμο να περνάει. Μετά το Brexit δεν υπάρχει πλέον αυτή η υποχρέωση της Γαλλίας. Η Μεγάλη Βρετανία θα πρέπει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα μόνη της. Δεν υπάρχει κάποια υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Γαλλίας. Αυτό πρέπει να το έχουν κατά νου όσοι είναι υπέρ του Brexit. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Brock. Now, Mr. Ο κύριος Φερχόφστατ, ευχαριστούμε τον κύριο Μπρόκ. Ε, αν ακούσει κανείς τον κύριο Μπρόκ θα θεωρήσει ότι η ε, Επιτροπή σας ε, ασχολείται με τα πάντα, ακόμα και, ε, με, την, τη συμφωνία του Τουκέ. Ακούστηκε πολλές φορές ο όρος τρίτη χώρα και πολλοί από τους Βρετανούς συναδέλφους στενοχωρήθηκαν. Δικαίως, αλλά δεν είναι δική μας επιλογή να, να, το, να χρησιμοποιούμε τον όρο αυτό. Η δική σας επιλογή είναι. Αν ας πούμε εσείς μας πείτε ότι δεν είναι δυνατή η ελευθερία κίνησης, τότε προφανώς δεν θα είναι δυνατή και μια συμφωνία τύπου Νορβηγίας. Αν μας πείτε ότι δεν μπορεί να υπάρχει εποπτεία από το δικαστήριο, τότε δεν μπορούμε να έχουμε μια συμφωνία τύπου Ουκρανίας, γιατί υπάρχει εποπτεία από το δικαστήριο. Όταν η Βρετανία λέει ότι θέλουμε να έχουμε τη δική μας κυριαρχία και τους δικούς μας κανόνες για τις εμπορικές συμφωνίες, τότε δεν είναι δυνατόν να υπάρξει τελωνιακή σύνδεση και συμφωνία. Ο λόγος για τον οποίο το συζητούμε δεν είναι επειδή εμείς το διαλέξαμε είναι επειδή εσείς το διαλέξατε. Οι δικές σας κόκκινες γραμμές είναι αυτές που μας μεταφέρουν από την πλήρη, από το πλήρως μέλος σε μια συμφωνία τάδε που δεν είναι δυνατή, σε μια τελωνιακή συμφωνία που δεν είναι δυνατή κτλ. κτλ, κτλ. Και σήμερα, σήμερα μιλούμε για μια συμφωνία με μια τρίτη χώρα. Αυτές είναι οι κόκκινες γραμμές οι δικές σας που μας δείχνουν τι έχουμε επιτάπητος για να διαπραγματευτούμε. Δεν είναι δική μας επιλογή, ούτε επιθυμία των 27 να πούνε εμεί θέλουμε αυτό ή θέλουμε το άλλο. Το μόνο που δεν μπορεί να γίνει είναι να δημιουργήσουμε μια κατάσταση και για τα περιβαλλοντικά πρότυπα που να είναι ίδια για τα πάντα. Οικονομικές υπηρεσίες, ακόμη και αν σας έλεγα για τις οικονομικές υπηρεσίες, το ίδιο είναι. Που ουσιαστικά στο τέλος θα υπονομεύει την Ένωση. Τώρα, α πούμε, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μία χώρα από τις 28. Όταν μιλούμε για θέματα περιβαλλοντικών προτύπων, είσαστε στην Κομισιόν, είσαστε στο Κοινοβούλιο, είσαστε μέλη στι διάφορες ε, υπηρεσίε, στο Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων και συνεργάζεστε με τα άλλα 27 κράτη και μαζί από κοινού καταλήγουμε σε μια συμφωνία. Μπορεί καμιά φορά να υπάρχει μια ε, ε, μειοψηφία που μπορεί να μπλοκάρει αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Αυτό που δεν μπορούμε να επιτρέψουμε είναι αυτό το σύστημα να αντικατασταθεί από ένα διμερές σύστημα για το οποίο για κάθε περιβαλλοντικό πρότυπο έχουμε 27, ε, Συμφωνία Ευρωπαϊκή 27 που θα την διαπραγματευτούμε με τον Ηνωμένο Βασίλειο μόνο του. Ε, τότε ας την παρατήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί δίνει ένα μήνυμα σε όλους, φύγετε και ουσιαστικά θα κερδίσετε και δύναμη, θα κερδίσετε κυριαρχία και για οποιοδήποτε πρότυπο, για υπηρεσίε υγεία, για περιβαλλοντικά, οποιαδήποτε συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση 27, τη Ευρω... μελλοντική Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή, και του Ηνωμένου Βασιλείου θα έχετε κι εσεί μια παρόμοια κατάσταση. Όχι, δεν θα είναι έτσι. Ούτε για τι οικονομικέ χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίε, ούτε για το περιβάλλον σε κανέναν τομέα τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα το επιτρέψουμε, γιατί αυτό υπονομεύει την Ένωση και δημιουργεί ένα νέο σύστημα όπου μια χώρα είναι μέρο των 28 και μετά το ε, αντικαθιστά αυτό με ένα διμερέ σύστημα και αυτοί που φεύγουν κερδίζουν και κάνουν εξίσου ικανέ συμφωνίες με την ε, Ευρώπη των 27. Το, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει την ε, δυνατότητα να καθορίσει τις, ε, τους κανόνες του. Θα υπάρχουν, θα κάνουμε βεβαίως διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περίοδου με τον Ηνωμένο Βασίλειο. Προφανώς θα υπάρξει στο μέλλον σύστημα διαμεσολάβησης ή διαιτησίας για τις μελλοντικέ σχέσεις αν υπάρχουν ας πούμε διαφορές. Αυτό που σίγουρα δεν θα κάνουμε ποτέ είναι να υπονομεύσουμε την αρχή των 27 να αποφασίζουν για αυτά τα πρότυπα και να τα επιβάλλουν αυτά τα πρότυπα. Οι διαβουλεύσεις λοιπόν για την μεταβατική περίοδο ναι, Δια, για το μέλλον ναι, όλα αυτά θα είναι δυνατά. Αλλά όχι η δυνατότητα και η αυτονομία των 27 ε, ε, να αποφασίζουν, ε, να υπονομεύεται η δυνατότητα αυτή των 27 να αποφασίζουν. Θα υπάρχουν διαβουλεύσεις, αλλά δεν μπορούμε να δώσουμε εξωτερική εργολαβία σε άλλους για να καθορίσουν πώς θα είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, οι σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί ουσιαστικά έτσι εκχωρούμε δική μας ε, αρμοδιότητα και δική μας εξουσία σε άλλους. Και αυτό δεν θα γίνει. Όπως και ο Έλμαρ Μπροκ. Και εγώ ακούω ότι λέμε ναι αλλά θέλουμε όλα τα, να μείνουν όπως είναι. Μα δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Είναι αδύνατο. Και δεν μπορούμε αυτό να το χρησιμοποιούμε όλη αυτή την συζήτηση για να υπονομεύουμε την ε, εξουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, δεν θα επιτρέψουμε ποτέ τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ε, αποδυναμωθούν. Αυτό είναι το κατώτατο όριο. Τα δικά μας ε, πρότυπα θα είναι το κατώτατο όριο, όπως κάνουμε πάντα όταν μιλούμε για σχέσεις με άλλη χώρα. Αυτά θα παραμείνουν απαράλλαχτα. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπονομευθούν τα δικά μας πρότυπα. Και αυτό δεν πρόκειται να γίνει ε, προσπάθεια για να επιδεινώσουμε οι μεν τους δε. Μπορούμε να έχουμε και άλλα πρότυπα. Ναι, μπορούμε ή για άλλους τομείς. Ε, για πρότυπα εργασία, ας πούμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει. Τρίτο στοιχείο. Πώς θα τα εφαρμόσουμε όλα αυτά. Έχουμε σύστημα συγκεκριμένο, όπως σε όλες τις συμφωνίες με τις τρίτες χώρες. Ένα συγκεκριμένο σύστημα διαιτησίας αλλά όταν έχει να κάνει με την ερμηνεία τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, δεν, θα γίνει, δεν θα γίνει η ερμηνεία από, την, από τη Διευθυνσία. Το Δικαστήριο του Ευρωπαϊκό θα κάνει την ερμηνεία όταν μιλούμε για την ερμηνεία τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Μόνο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα έχει την αρμοδιότητα και την εξουσία να το κάνει. Και αυτό είναι βεβαίω ανεξάρτητα από τη διαιτησία. Διαιτησία, α πούμε, μπορεί να γίνει όταν υπάρξει ερμηνεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διαιτησία θα σε στείλει στο δικαστήριο. Δεν θα κάνει η ε, δεν θα αναλάβει η εργολαβία την, η διαιτησία την ερμηνεία τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Μετά, για τη μετάβαση. Κυρία Γκέρλινγκ η μετάβαση είναι κομμάτι της απόσυρσης, της αποχώρησης, δεν είναι ξεχωριστό κομμάτι. Είναι κομμάτι της αποχώρησης, άρθρο 50. Αυτό είναι ένας από τους λόγους που αυτή η μετάβαση δεν μπορεί να κρατήσει 10 χρόνια. Γιατί μετά δεν είναι μετάβαση πια. Ούτε μετά μπορούμε να την αποτελέσει κομμάτι της αποχώρησης. Είναι αποχώρηση, είναι κομμάτι της αποχώρησης που σημαίνει ότι είναι περιορισμένη σε χρόνο. Ο κύριος Μπαρνιέ λέει μέχρι το 2020. Και εμείς λέμε, εντάξει, ίσως και λίγο παραπάνω, άντε το πολύ τρία χρόνια, αλλά θα είναι κομμάτι της αποχώρησης. Οπότε, όταν υπάρξει συμφωνία εδώ στο Κοινοβούλιο τον Οκτώβριο του τρέχοντος, θα είναι η αποχώρηση μέσω του άρθρου 50, συν την ε, μεταβατική περίοδο, συν ένα παράρτημα κατά πάσα πιθανότητα, που θα είναι μια πολιτική δήλωση για τις μελλοντικέ σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο. Πάω λίγο γρήγορα για τα διάφορα σχόλια που έγιναν. Νομίζω ότι είναι απολύτως σαφές ότι πρέπει να βρεθούν λύσεις. Τις, ε, το ξέρουμε, ας πούμε, για την έρευνα, για την Ευρατόμ, ε, Έχουμε πολλά παραδείγματα για το πώς δουλεύουν όλα αυτά με τρίτες χώρες και έχουμε ε, και τη δυνατότητα να ε, χρησιμοποιήσουμε τέτοιους μορφοτύπους και στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου. Τελευταίο σχόλιο για τον κύριο Φλάναγκαν που είπε αν είσαστε, ότι εσείς είστε ο καλός α, ε, ε, ε, διαπραγματευτής γιατί είσαστε, καλός, γιατί είσαστε φε, και ο Σούμαν φεντεραλιστής ήταν και ο Τσόρτσιλ νομίζω ότι φεντεραλιστής ήταν αλλά εν πάση περιπτώσει δεν νομίζω ότι αυτό θα αποτελέσει πρόβλημα. Είπα ότι κάποιες χώρες θα είναι οι νάνοι του μελλοντικού κόσμου ο μόνος τρόπος για να το αποφύγουμε αυτό είναι να συνεργαζόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι ο Πόλαν Ρι Σπακ το είπε. Κάποιοι είναι, όλοι μας είμαστε νάνοι. Κάποιοι το ξέρουν, κάποιοι δεν έχουν τις γνώσεις αρκετά για να το ξέρουν. Έτσι έχει η κατάσταση. Νομίζω λοιπόν ότι σημείο κλειδί είναι Πρόεδρε, αν γίνεται για τα πέντε ερωτήματα που έθεσα να λάβουμε απαντήσεις, να μας πείτε τις απόψεις σας, έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε τις ε, απόψεις και, εσείς, και τις δικές σας για το ε, ψήφισμα. Ε, το ψήφισμα δεν, είναι, δεν έχει καταγραφεί ακόμα, θα γραφεί τέλος Φεβρουαρίου μόλις θα λάβουμε από την Επιτροπή σας τις προτάσεις σας και τα σχόλιά σας για να, μπει στο, να μπουν στο κεφάλαιο που θα αφορά στο περιβάλλον. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Um, we invite you to come again. Θα σας ξανακαλέσουμε όταν θα ε, έχουν γίνει νέα βήματα ως προς το Brexit. Σας ευχαριστώ πολύ και θα τα πούμε την επόμενη φορά.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 Αγαπητοί συνάδελφοι, αν έχετε έτοιμες ε, τις ε, κάρτες σας, Then we start the voting. μπορούμε να αρχίσουμε με τις ψηφοφορίες. Πριν θα ήθελα να χαιρετήσω τους φοιτητές που κάλεσε ο κύριος ε, Φλόρενς από το Πανεπιστήμιο του Πρέβε μαζί με τον καθηγητή Σίγκιν. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν. Το πρώτο θέμα για ψηφοφορία είναι οι κοινές προσπάθειες στο κατάλογο effort sharing. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, άρχεται η ψηφοφορία. ένας υπεράριθμος από το ΕΛΚ. Εντάξει. Πέρας. Και εγκρίθηκε. Συγχαρητήρια. Τώρα μπορούμε να ψηφίσουμε για το Λουλουσιεφ. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ένας υπεράριθμος από το L και πάλι. Πάλι ένας υπεράριθμος. Μπορούμε να το λύσουμε αυτό για να ε, το λύσουμε. Μπορεί κάποιος να αποσύρει την κάρτα του από το ΕΛΚ. Πέρας και εγκρίνεται συγχαρητήρια. Η επόμενη είναι μία προφερική ερώτηση προς την Επιτροπή για τον εμβολιασμό και τη μείωση των ποσοστών εμβολιασμού, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας και εγκρίνεται. Επίσης, ε, προφορική ερώτηση προς το Συμβούλιο, ίδιο ερώτημα, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Next, uh, next uh, vote is um, on the draft report εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα που προέρχονται από τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα. 15 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. Ενενήντα τέσσερα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ενενήντα έξι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ενενήντα επτά υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ενενήντα οκτώ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 99 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 102 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 103 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 105 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 106. Όχι. Καταπίπτει. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τραν 16 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Και πέρας. Και εγκρίνεται. Εκατόν δεκαοκτώ. Εκατόν δεκαοκτώ υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 119 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 120 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 121 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 122 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 123 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 124 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε την 124 άρχεται η ψηφοφορία 124 πέρας εγκρίνεται 125 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 127. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 128. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τραν 19. Υπέρ. Κατά Ελέγχουμε την τραν 19. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται συμβαστική 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 131 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 137 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 138 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 8 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 23, 152 και 153 είναι επανομοιότυπες υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 154 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 24 και τραν 24 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 155 και τραν 25. 25 και 26 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 156 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 157 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 158 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 159 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 160 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 161 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 162 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική 11 υπέρ κατά εγκρίνεται η συμβιβαστική. 173 και 174 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. 175 υπέρ. Κατά αποχές ελέγχουμε την 175. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 184 υπέρ. Κατά. Αποχές ελέγχουμε την 184. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. 185 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 186 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 187 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 188 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τραν 1 υπέρ. Κατά. Αποχές Ποιο είναι υπέρ, υπέρ παρακαλώ. Εγκρίνεται. Τραν 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 38 υπέρ. Θέλετε να ελέγξουμε τη 37. Άρχεται η ψηφοφορία. πέρας απορρίπτεται. 38 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 39 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 41 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τραν 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 44 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 46 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 47 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 53 υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται. 55 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 56 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 57 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 58 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τρανέντεκα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 8 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε την 8 Πέρας. Εγκρίνεται. Εννέα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν βλέπω το ΕΛΚ τι κάνει. Εννέα υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε την εννέα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 70 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 71 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 77 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 79 και 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 87 όχι, με συγχωρείτε, συμβαστική 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 87 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τι θέλετε να ελέγξουμε. Ελέγχουμε. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 88, 89, 90, 14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται 91 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται τραν 15 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 92 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 93 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται η έκθεση όπως έχει τροποποιηθεί, υπέρ... α, ηλεκτρονικά με συγχωρείτε, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας και εγκρίνεται. Τώρα θα ψηφίσουμε για την εντολή για να αρχίσουν οι διαθεσμικές διαπραγματεύσεις. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρας. Πέρας. Εγκρίνεται η εντολή. Χωρίς ε, μεγάλη πλειοψηφία. Next one is... Uh, Επόμενο σημείο. Έκθεση της κυρίας Αγιούσο. Ψηφίζουμε για την επισήμανση των ακολούχων ποτών. Τροπολογία 159. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε παρακαλώ. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, αρχιτεί η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την 159. Πρώτη είναι, αλλά ήταν μισή-μισή η υπέρ και η κατά. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2.160 άγκρι 12. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 161 υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. 3. Άγκρι 13 και... Α, αυτές τις δύο μόνο. 3 και 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Άγκρι 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 162. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 163 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 164 υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 165. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 166. 167. 168 και εξή 169 και 170. Όχι, σταματάμε εδώ. Λοιπόν, 167 και 168. Η 166 αποσύρεται. Ποιος είναι υπέρ 167-168? Κανείς. Κατά. Απορρίπτονται. 167 ε, και 168 ψηφίσαμε, έτσι. Λοιπόν, πάμε στην 169 και 170. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Άγκρι 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 171. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 173. 172-173-17 ε, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. Άκρη 18 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 174 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 175 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 21 και είναι τα 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 177 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ποιος το είπε αυτό. Λοιπόν, το ελέγχουμε ηλεκτρονικά, ψηφίζουμε. Μπορεί να έχετε και δίκιο. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 178 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 179 υπέρ. Κατά. Αποχές. 179 παρακαλώ ξανά. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 180 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 181 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 5 και άγκρι 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 182 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 183 και 184 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εντάξει, να το ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 183 και 184. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνονται. Τρόπολογια 6 και άγκρι 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 185, 186. Υπέρ. Κατά αποχές ελέγχουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ Αρχιτή ψηφοφορία και πέρα ψηφοφορίας εγκρίνονται 187 και άγκρι 24 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές δεν ψηφίσατε 187 και άγκρι 24 παρακαλώ ψηλά τα χέρια σας υπέρ, κατά, αποχές. Να το ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνονται. Πακέτο για την ε, περιεκτικότητα στη σάκχαρα. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 190, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 191 υπέρ «191 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται». «192 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται». «194 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται». «195 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Διακόσια 23, 24, 25 υπέρ κατά αποχές Ελέγχουμε. 2.22, 2.23, 2.24 και 2.25. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτονται. 2.21 υπέρ. Κατά αποχές, απορρίπτεται. 2.26 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2.27 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2.28 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2.29 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2.30 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2.31 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Άγκρι, 13, άγκρι 31, συγγνώμη, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ε, στην τροπολογία 8, καταπίπτει. Άγκρι 32, υπέρ, κατά, αποχές, να το ελέγξουμε παρακαλώ. Άγκρι 32. Πέρας, απορρίπτεται. Άγκρι 33, υπέρ, κατά, Αποχές. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άγκρι 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Μπλοκ 232, 233, τα 9 και Άγκρι 35 από κοινού. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 234 μέχρι την 2.37 είναι τα 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 2.38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται άγκρι 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 2.41 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 2.43 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 2.44 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 2.45 υπέρ. Κατά αποχές απο... εγκρίνεται. 2.47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 38 και 2.48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.49 υπέρ κατά αποχές εγ... απορρίπτεται. 2.50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.52 υπέρ κατά Αποχές. Απορρίπτεται. 2.53. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.54. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.55. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.56. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.58. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.57. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.59. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.60 και 2.61 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές δεν είδα το άλλο αυτή τη φορά τι ψήφισε. 2.60 και 2.61 παρακαλώ, υπέρ. Κατά. Αποχές να το ελέγξουμε. Παρόλο που είδα τελικά τι ψηφίσατε, δεν κατάλαβα. Άρχιδη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 2,62 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2,64 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2,63 και άγκρι 39 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 268 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 266 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 275, 276, 77 και 78 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 2,74 υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Άρχιδη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 2,79 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 283. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 302. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 303 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 304 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 305 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 είναι τα 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 52 και είναι τα 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3.12 και άγκρι 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Άγκρι 57 και είναι τα 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 3.14 και άγκρι 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Κατά 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Κατά υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. είπέρ. υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 3-19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 321 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 322 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 323 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 324 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 325 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 326 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 327 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. Τροπολογία 14 και είναι 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 328 και 329. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ποιος είναι κατά. Εγκρίνεται. 330. Υπέρ. Α, συγγνώμη. Καταπίπτει. Συμβαστική 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3.36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 3.37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 3.38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 3.39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 3.40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 3.41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 3.42 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. Είναι τα 25 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 16. 343 και είναι τα 26 υπέρ. Κατά αποχές. Α, εγκρίνονται. 17. 344 είναι τα 27 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνονται. 18 είναι τα 3.45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 19.346 ίντα 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Άγκρι 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ίντα 30 υπέρ κατά αποχές. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την ίντα 30 άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας Απορρίπτεται. 3.47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3.48 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Άγκρι 62 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν κατάλαβα. Ποιος είναι υπέρ για το 62. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 20, 32 και 349 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 350 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Άγκρι 63 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 21 είναι 33 και 351 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Είναι 34 και άγκρι 64 υπέρ. Κατά αποχές, εγκρίνονται. Συμβαστική 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Άγκρι 66 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 357 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 358 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άγκρι 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 359 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 23 υπέρ, είναι τα 37 και, και τίποτα άλλο. Ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 360 υπέρ κατά Αποχές. Απορρίπτεται. τα 38. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 371. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 372 υπέρ καταπίπτει. 373 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 70 υπέρ <clears throat> κατά αποχές εγκρίνεται. 374 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 375 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 376 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 18 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 393 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 31 και άγκρι 74 υπέρ. Κατά. Αποχές. εγκρίνονται. 394 υπέρ. Κατά. αποχέ, Απορρίπτεται. 396 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 397 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 397. Ωραία. Την ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας πληροφορία. Απορρίπτεται. Θέλετε να ελέγξουμε και την 396. Ωραία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 396, άρχεται η ψηφοφορία. And it's closed. And it is Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρι, όχι καταπίπτει. Πάμε στην 401, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 402, 403, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Όλα αυτά θα τα ψηφίσουμε. 402-403. Άρχεται η ψηφοφορία. Μου κάνει και θόρυβο. Πέρας. Εγκρίνεται, ζητώ συγγνώμη. Ωραία. Μετά δεν ψηφίζουμε για τα υπόλοιπα, αλλά σας ευχαριστώ για την πρόταση. Μα εγκρίθηκε. Αχ, όχι αυτό. Ωραία. 405 υπέρ. Κατά. 405 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να την επαληθεύσουμε. Ε, δεν βλέπω. Εγκρίνεται. Άρχεται ε, και πέρας. 404 υπέρ. Α, καταπίπτει. Μάλιστα, τροπολογία 33 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 406 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 407 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 409 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 408 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 76 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 77 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 410 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 411 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άγκρι 78 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άγκρι 79 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άγριο 80 υπέρ. Κατά. Αποχές. 412 4-12 υπέρ. Κατά. Αποχές. 413 4-13 υπέρ. Κατά. Αποχές. 414 και 415 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τεχνικό συμβιβασμός παράρτημα 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Σελίδα 38. Ψηφίζουμε την 418 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 421 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 4.22 υπέρ. Κατά. Αποχές να την επαληθεύσουμε. 4.22. Α, υπήρχε μια καθυστέρηση μάλιστα, εγκρίνεται. 4.23 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Να την επαληθεύσουμε. 4.23. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 4, 24 υπέρ κατά αποχές. Ε, δεν μπορώ να δω. 4, 24 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 4, 26 υπέρ. Κατά. Ο κύριος Ντάνς κάνει έτσι. Ε, τι να πω. 4.26 υπέρ. Ευχαριστώ. Εγκρίνεται. 4.28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4, 32, 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 4.37 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 4. Να, μάλιστα, συμβαστική 19 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 4.40, πρώτο μέρος υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ναι, να επαληθεύσουμε το πρώτο μέρος της 4.40, ε, άρχεται η ψηφοφορία, αλλά το ΕΛΚ και οι σοσιαλδημοκράτες ψηφίζουν το ίδιο. Εγκρίνεται. Άγκρι 90 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4.42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 4.42 ναι, μπορώ να σα ξαναρωτήσω αν θέλετε. 4.42 όλα. Α, δείξτε. Ε, τα χεράκια, σκόστε τα χεράκια. Δεν έχω πρόβλημα εγώ με καμία τροπολογία. ορίστε λοιπόν, εγκρίνεται. Ζητώ συγγνώμη από τον κύριο Πιέκα. Αλλά δεν είχατε σηκώσει, δεν έχει σηκώσει κάνει το χέρι εκτό από εσά. Συμβαστική 20 υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. 4.48 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 4.41 και εγκρίνεται. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4.50 υπέρ. Κατά. Να το επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. και πέρας. Εγκρίνεται. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 454 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 459 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 460 και 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 462 και 463 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 464 και 465 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 466 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 467 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 468 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 469 υπέρ κατά αποχές απολύτεται. Συμβαστική 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4,72 υπέρ. Κατά αποχές να την επαληθεύσουμε. Πέρας απορρίπτεται. σε διαβαστική 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πέντε 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5-17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρε 100 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5, 18 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 71 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 101 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 5-20 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 75 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 77 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 79 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Θέλετε να ψηφίσουμε, να τις ψηφίσουμε όλες μαζί μέχρι το 88. 81-88. Λοιπόν, 81-88 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Απορρίπτονται όλες. 96 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Αγκρία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 89 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 90 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 91 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά. 92 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 93 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 94 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 95 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 97 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 98 υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι εγκρίνεται. Ας το επαληθεύσουμε. 98. Άρχεται η ψηφοφορία. Και πέρασε. Και απορρίπτεται. Άγκρι 2. Υπέρ κατά αποχές ε, γκρίνεται. 99 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 100 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 108 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 109 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 101 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 3 υπέρ. Κατά. Αποχές, να το επαληθεύσουμε. Άγκρι 3 λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Και πέρας. Και εγκρίνεται. 102 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 120 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 103 υπέρ και 104 υπέρ κατά αποχές να την επαληθεύσουμε 103 και 104 Απορρίπτεται. 105 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και προτείνω ξανά όλες μαζί από την 106 μέχρι την 115 αν είναι δυνατόν στον κατάλογο ψηφοφοριών. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, είπατε όχι. Ο κύριος Πετιτσίνη, μάλιστα, 106 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 107 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 110 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 111 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 112 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 113 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 114 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 115 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 117 υπέρ και 118 και 119 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 116 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 121 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 122 υπέρ Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 123 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 124 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 125 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 132 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 133 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Άκρη 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 135 και άγκρι 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 137 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 138 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Είναι τα 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 8 υπέρ. Συγγνώμη, μάλλον καταπίπτει. Άγκρι 10 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 140 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 141 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 142 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 143 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 144 υπέρ κατά να την επαληθεύσουμε άρχεται η ψηφοφορία και πέρασε. και εγκρίνεται Συμβαστική 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 43 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 154 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 155 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 156 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 157 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 158 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, τελική ψηφοφορία ηλεκτρονική, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται. Μπράβο. Συγχαρητήρια κυρία Γιούζο. Έχουμε ακόμα πόσες εκθέσεις. Έχουμε 7 8 ψηφοφορίες ακόμα. Για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου ε, κυρία Γιάτεμακη, συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε την 16 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε την 18 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Θέλετε να ελέγξουμε, ελέγχουμε. Ελέγχουμε την 30. 1. Πέρας. Απορρίπτεται πράγματι. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 41 μέχρι και 45 είναι παρόμοιες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 46 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε την 46 άρχεται η ψηφοφορία πέρας και εγκρίνεται 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Όχι, με συγχωρείτε, απορρίπτεται. 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 54 υπέρ κατά αποχές ε, ελέγχουμε την 54 εγκρίνεται ζητώ συγγνώμη εγκρίνεται 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 58 όχι 65 και 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 66 70 74 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 68 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 71 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 82 υπέρ. Κατά όχι, όχι, έκανα λάθος, με συγχωρείτε, έχω κάνει ένα μεγάλο λάθος, με μπερδεύουν τα χρώματα. Συμβαστική 5, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 82, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 83, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 85, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 86, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται.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 Επόμενο θέμα. Okay. Um, so, a European strategy... Ευρωπαϊκή στρατηγική για συνεργατικά και ευφυή συστήματα μεταφορών. 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ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 38 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 39 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 40 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 40 43. Υπέρ. Φαίνεται ότι ψηφίσαμε τη 42. Εγκρίθηκε. 43 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 45 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 46 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 48 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά η οποία και άρχεται.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 αποχές ε, ελέγχουμε για το δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται. 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρι... Α, ε, ελέγχουμε μάλλον.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 κατά αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Α, ας το ξανακάνουμε. 20 υπέρ. Εγκρίνεται, εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 22 υπέρ κατά αποχές Ελέγχουμε την 22. Άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 24 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα έχουμε τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά, η οποία και αρχίζει. Και πέρας εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Τώρα, απαλλαγή. Αρχίζουμε τις απαλλαγές. Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρώτα.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 Πέρας και εγκρίνεται. Ψηφίζουμε για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων 1 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 2 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 5 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 με μια προφορική. Δέχεστε την προφορική. Τροπολογία. Ωραία. Ψηφίζουμε λοιπόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 9. Που έχει επίσης προφορική. τη δέχεστε. Ωραία, ψηφίζουμε την 9 υπέρ κατά αποχές. Ας ελέγξουμε την 9 με την προφορική. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας και απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Απαλλαγή για την ΕΦΣΑ. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 2. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 10 υπέρ Α, δεν ψηφίσαμε την 8. 8, τροπολογία 8 υπέρ, εγκρίνεται, 10 υπέρ, κατά, ελέγχουμε την 10, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας και εγκρίνεται 9 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά άρχεται. Πέρας και εγκρίνεται. Τώρα περνάμε στην απαλλαγή για το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων. Ένα υπέρ κατά αποχές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 Κατά. Ελέγχουμε, ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για την 1. Πέρας. Απορρίπτεται. 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 3. Ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 6. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά η οποία και αρχίζει. Πέρας και εγκρίνεται. Ε, απαλλαγή έκα 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τρία υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τέσσερα υπέρ κατά αποχές ε, ελέγχουμε την 4 άρχεται η ψηφοφορία πέρας και απορρίπτεται 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία Πέρας και εγκρίνεται. Και τελειώσαμε με τις ψηφοφορίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία σας και την κατανόηση. Όπως ξέρετε, η κυρία Μπιενκόφσκα ε, τη ζητήθηκε μάλλον να απαντήσει γραπτός. Άρα τελειώνουμε με τη σημερινή μας συνεδρίαση.